τη χθεσινή συνεδρίαση και τα κείμενα που υιοθετήθηκαν. στη διάθεσή σα και ρωτώ αν υπάρχουν σχόλια. Εάν όχι, εγκρίνονται τα πρακτικά και σας ευχαριστώ.